Περνάμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης. Την εκλογή δηλαδή αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω λάβει τα εξής ονόματα υποψηφίων. Ρομπέρτα Αντζελίλη. Μπέλ. Καμίνσκι Μίχαου Τόμας. Κοχ Μέριν Σιλβάνα. Κράτσα Τσαγκαροπόλου. Rodi Lambrinidis Stavros Macmillan Scott Edward Martinez Martinez Miguel Angel Pitella Giovanni Rod Berend Dagmar Rouczek Libor Schmidt Paul Vidal Quadras Alejo Wallis Diana Wieland Reiner. Έχουμε περισσότερους δηλαδή από 14 υποψηφίους ενώ είναι 14 οι αντιπρόεδροι οπότε θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία στον πρώτο γύρο της ε, ψηφοφορίας. Οι δε καταμετρητές των ψήφων θα είναι ακριβώς οι ίδιοι που ήταν και για την ε, εκλογή του Προέδρου, οπότε σας παρακαλώ να μετακινηθείτε στις ε, κάλπες και να θυμάστε ότι θα ψηφίσετε τελευταίοι. Επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού, επειδή έχουμε περισσότερους υποψηφίους αποθέσεις, θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία. Διαβάζω το ε, σχετικό άρθρο. Όλοι χρησιμοποιούν μόνο μία κάρτα και επιλέγουν το άτομο το οποίο θέλουν να ε, ψηφίσουν. Σας παρακαλώ καθίστε γιατί διαβάζω άρθρα από τον ε, κανονισμό και το τι πρέπει να γίνει τα επόμενα 20 λεπτά. Στον, ε, στον πρώτο γύρο έχουμε 14 θέσεις. Όσοι υποψήφοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων θα εκλεγούν. Εάν ο αριθμός ε, αυτός και πάλι υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος. Εάν περάσουμε σε τρίτο γύρο αρκεί απλή πλειοψηφία. Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω πως έχετε λάβει ψηφοδέλτια και φακέλου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να χρησιμοποιήσετε μόνο τα ψηφοδέλτια τα οποία έχετε λάβει. Θα επιλέξετε το όνομα του υποψηφίου που θέλετε να ψηφίσετε, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχουν 14 θέσεις Σφοδέλτια δε τα οποία έχουν παραπάνω από 14 σταυρούς θεωρούνται άκυρα. Εάν θέλετε να διορθώσετε κάτι θα ζητήσετε από έναν κλητήρα ένα νέο ψηφοδέλτιο, το παλιό ψηφοδέλτιο θα καταστραφεί, οποιοδήποτε άλλο διακριτικό γνώρισμα ή χαρακτηριστικό ή πάνω από 14 σταυροί, όλα αυτά καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. Όταν ε, ψηφίσετε, τοποθείτε το ψηφοδέλτιό σας μέσα στον φάκελο. Κύριοι και κυρίες, αγαπητοί συνάδελφοι, κηρύσω την έναρξη της ψηφοφορίας. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει ε, κάποια ελάχιστη απέτηση για την ψηφοφορία, ελάχιστος αριθμός σταυρών. Όχι, ε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή, κύριε Σάιερ. question. Σας ευχαριστώ για την ερωτησή σας. Δεν υπάρχει κάποιος ελάχιστος αριθμός. Μπορεί να είναι μόνο ένας ή δύο, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας.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 is last moment for voting. Τελευταία σας ευκαιρία για να ψηφίσετε είναι τώρα. Some of you are moving very quickly. I understand they want to take part in election. Κάποιοι από εσάς ε, κινούνται έτσι ώστε να πάρουν μέρος τελικά στην ψηφοφορία. Ε, I am asking you second time, is anybody too ready to take part in the election? Θέλει κάποιος άλλος να ψηφίσει. Σας ρωτάω δεύτερη, σας ρωτάω και μια τρίτη φορά. Well, ladies and gentlemen. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. τη Πέρας της ψηφοφορίας. Επαναλαμβάνω πέρας. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τους καταμετρητές ψήφων να πάνε στο δωμάτιο R01101 για να κάνουν την καταμέτρηση. Διακόπτεται η συνεδρίαση και θα επαναληφθεί όταν ακούσετε το κουδούνι. Σε μία ώρα τουλάχιστον περίπου. Ίσως και 45 λεπτά, αλλά οπωσδήποτε όχι παραπάνω από μία ώρα. Διακόπτεται η συνεδρίαση.